μου ζήτησε να σας ενημερώσω για την ε, ίδρυση της, ε, της, την επανίδρυση της ε, πολιτικής ομάδας EFDD από την 20η Οκτωβρίου του 2014 46 βουλευτές απαρτίζουν την ομάδα Μέσης Δημοκρατίας και Ελευθερίας το άρθρο 32 ε, του εσωτερικού κανονισμού εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Αυτή είναι η ενημέρωση ε, εκ μέρους του Πρόεδρου. Ε, Ευχαριστώ. Φαντάζομαι επιδοκιμάσετε τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύω στην Ολομέλη.